Good morning. Καλημέρα σε όλους σας. Ok. Apriamo la seduta Συνεχίζει η συνεδρίαση της Επιτροπής. Με πληροφορίες καταρχήν σχετικά με το τι αποφάσει πήραν οι, οι συντονιστές χθες. Η πιο σημαντική πληροφορία είναι ότι ουσιαστικά αποφασίσαμε να κλείσουμε το pipeline. Σας εξηγώ τι εννοώ. Είχαμε πάρει μια πρόταση της Κομισιόν, πρόταση οδηγίας, για το τι ισχύει για τα πλοία που μπαίνουν ή βγαίνουν από τα κοινοτικά λιμάνια. Ένα νομοθετήμα. Αν έπρεπε να ορίσουμε εισηγητή, θα αρχίζαμε να εργαζόμαστε τώρα, αλλά δεν θα προλαβαίναμε να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία μέχρι τον Ιούνιο. Και ουσιαστικά η δουλειά θα ήταν περιττή. Γι' αυτό αποφασίσαμε να μην ορίσουμε εισηγητή, να μην δώσουμε συνέχεια στην πρώτη αλλαγή της οδηγίας και σημειώστε το εξής. Θα στείλω μια επιστολή στον Επίτροπο Ταγιάννη θα του πούμε ότι λυπούμαστε που ήρθε τόσο αργά αυτή η πρόταση οδηγία. Αν έχει γίνει πιο πριν θα μπορούσαμε να ορίσουμε και κλπ. Οπότε, εκτός αν υπάρχουν άκρες εξαιρέσεις, θεωρούμε ότι είναι περιττό να μας αναφέρουν αλλαγές στην νομοθεσία οτιδήποτε στα οποία θα πρέπει να δοθεί συνέχεια, ενώ δεν είναι δυνατόν να γίνει. Στου επόμενου μήνε λοιπόν, θα του πω, θα προσπαθήσουμε να κλείσουμε όσα θέματα έχουμε ανοιχτά στο pipeline, χωρίς να τα τροφοδοτούμε με νέο υλικό, νέες προτάσεις. Εξαίρεση θα σήμαινε θα έπρεπε να ζητήσουμε από την ΓΚΟΕ, να αριστερά, να αριστερά, να ορίσει εισηγητή για τον προπολογισμό, άλλα για Μάρκο Πόλο κλπ. κλπ. Δηλαδή ουσιαστικά αυτό που θεωρούμε ότι είναι δυνατό να έρθει σε πέρας μέχρι τον Ιούνιο θα το κάνουμε. Ότι όμως υπάρχει κίνδυνος να είναι άχρηστη, περιττή δουλειά δεν θα το κάνουμε. Αυτό που εμείς θέλουμε να κάνουμε, όπως εκθέσεις πρωτοβουλίες, δεν μπορούμε να τις κάνουμε. Γι' αυτό που μας λένε να δουλέψουμε, ενώ είναι περιττή η εργασία αυτή, αυτή είναι η θέση μας όπως την περιέγραψα. Μεταξύ των εγγράφων που μας ήρθαν προς πληροφόρηση και προς ανάλυση υπάρχει και το σημείο 9 της χθεσινής ημερήσιας διάταξης, μια έκθεση για τη χρηματοδότηση για την ασφάλεια στην αεροπορία. Εξωτερική ασφάλεια. Θυμόσαστε στο πακέτο ε, συμβιβασμού στην αλλαγή του κανονισμού για την ασφάλεια. Είχαμε συνδέσει το θέμα αυτό με ένα αίτημά μας να κάνει πρόταση η Κομισιόν. Σωστά, η Κομισιόν ξεκινάει με ανακοίνωση ως εδώ καλά. Αλλά η μετριοφροσύνη της πρότασης αυτής, τη ανακοίνωση, μάλλον αυτής, και μία ανακοίνωση σημαίνει ότι δεν, σημαίνει δεν θα έχουμε πρόταση νομοθετική, σημαίνει ότι δεν τηρήθηκε η ανάληψη, η δέσμευση μάλλον που αναλήφθηκε από την Κομισιόν. Θα γράψουμε λοιπόν στον Επίτροπο Ταγιάννη και θα παραπονεθούμε για την καθυστέρηση αυτή και θα του θυμίσουμε την παλιά μας θέση, κλασική θέση, ότι το κόστος της ασφάλειας θα πρέπει να υποδιαιρεθεί έτσι ώστε να λαμβάνει υπόψη το συμφέρον του κάθε ταξιδιώτη και ταυτόχρονα την ανάγκη τα κράτη να φέρουν το βάρος της ασφάλειας. Ιδιαίτερα στην περίπτωση που θα έχουμε πιο αυστηρά μέτρα, most, more stringent. Κατά συνέπεια, επιστολή και για το θέμα αυτό. Μια άλλη επιστολή χθε επίσης εγκρίθηκε για το CIS. Έκθεση Κίρκοπ. Και εκεί περιμέναμε η Κομισιόν να μας δώσει μια εξήγηση, μια ερμηνεία για το Parrot Carrier. Για όλα τα άλλα σημειώσαμε με ενδιαφέρον ότι ο οργανισμός θα συνεργαστεί με το πρόγραμμα της ΟΛΕΦ κατά των απατών. Έχουμε το, την ε, έκθεση Σαβαρή για την κινητικότητα, όπου απαιτείται διαβούλευση με την Επιτροπή Περιφερειών Ελπίζουμε το κείμενο από τη μεριά τους να έρθει σχετικά σύντομα, πάντως δεν θα περιμένουμε. Εμείς θα κινηθούμε με το δικό μας ρυθμό για την κινητικότητα, σοβαρή. Για τον εισηγητή μας Ρόμπερτ Evans, η Επιτροπή Περιβάλλοντος ετοιμάζει μια προφορική ερώτηση για την διάλυση των πλοίων θα ζητήσουμε να πάρουμε και εμείς μέρος. Θα ζητήσουμε από τον συνάδελφο Evans να το κάνει αυτό για να υπάρχει και η θέση της Επιτροπής Μεταφορών. Με αυτά τελείωσα για τις χθεσινές αποφάσεις. Αν έχετε έρθει όλοι, μπορεί να αρχίσει η ψηφοφορία. Αρχίζουμε. Συγγνώμη. Ε, ένα τεστ. Ένα τεστ στην αρχή να δούμε αν τα μηχανήματα δεν βάλετε την κάρτα σας στον μηχάνημα και ψηφίζουμε.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 Έχουμε δύο σοσιαλιστές επιπλέον. Να ξαναδοκιμάσουμε άλλη μια φορά. Allora, possiamo rivotare per favore? Παρακαλώ να ξαναψηφίσουμε. Fine. Close the vote. Ok, ma questo I have to see this. How can I? Okay. Allora. Μάλιστα. Ψηφίζουμε. Συμφωνία μεταξύ Ένωσης και Δημοκρατίας Αρμενίας σχετικά με ορισμένε πτυχές των αεροπορικών υπηρεσιών. Τελική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Επέρτα la votazione τίποτα το τούτη. Ψηφίσετε όλοι πέρας. 45 υπέρ, μία εποχή Εγκρίνεται. Ο κύριος Πουσα. Κύριε Πρόεδρε, ε, πριν από την ε, ψηφοφορία σε ό,τι αφορά τη συμφωνία, την αεροπορική συμφωνία... Sí. Okay πριν από την ε, ψηφοφορία. σε ποια συμφωνία αναφέρεστε, ποια συμφωνία αναφέρεστε τώρα, ε, πείτε μας. Μεταξύ του Συμβουλίου και του Ισραήλ θέλω να κάνω μια δήλωση. No, there is... Ψηφίζουμε. Είμαστε σε ε, διαδικασία ψηφοφορίας, η δήλωση μετά, μετά, όχι τώρα. Είπαμε αλλά αρχίζει η ψηφοφορία. Διαφορετικά θα ξεκινήσει η συζήτηση και δεν τελειώνει ποτέ. Σέβομαι απόλυτα ό,τι θέλετε να πείτε, θα προσθεθεί στα πρακτικά η δήλωση, αλλά όχι τώρα. Θα πρέπει να έχει γίνει πριν από ένα μήνα ή μετά την ψηφοφορία. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Αν ψηφίσατε όλοι, πέρας, 49 παρόντες, 48 ψηφίζουν, 44 υπέρ, 2 κατά, 2 αποχές εγκρίνεται. Η δήλωση θα μπει στα πρακτικά και θα χρησιμοποιηθούν όπως πρέπει. Okay, allora, Τώρα αρχίζει η ψηφοφορία. Πρόταση οδηγίας προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για αλλαγή της ε, οδηγίας για την Ευρωβινιέτ Η ο Ελκα Ντράουι. Τροπολογία 159 Γελοβιεύσκη. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τον συμβιβασμό Α σε χωριστά τμήματα. Πρώτο τμήμα είναι το σύνολο με εξαίρεση παράγραφο 2. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, αλλά θα κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 50 παρόντες, 48 ψηφίζουν, 32 πέρα 16 κατά. Καμία αποχή. Το πρώτο τμήμα εγκρίθηκε του συμβαστικού α. Ερχόμαστε στο δεύτερο τμήμα. Είναι υπό 2 υπέρ κατά ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψηφίζουμε.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 αποχές εγκρίνεται το τρίτο τμήμα της υποπαραγράφου 5. Έχετε μπροστά σας φαντάζομαι τις ε, τροπολογίες, βλέπετε ποιες καταπίπτουν. Αν θέλετε μπορώ να σας διαβάζω ποιες καταπίπτουν. Ερχόμαστε στη συμβαστική, στο συμβασμό Β, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται καταπίπτει ερχόμαστε στο συμβαστικό γάμα 464-67 κατά πέσα Δεν υπάρχει συμβαστική C, Γ και αυτή έπεσε. Ερχόμαστε στο J, συμβαστική υπέρ, κατά, αποχές. Το J, J εγκρίνεται. Συμβαστική D, Δέλτα. Στο άρθρο 1, σημείο 4, άρθρο 9, παράγραφος 2, σε τμήματικά. Το πρώτο τμήμα που είναι όλος ο συμβασμός Δέλτα, με εξαίρεση συμπεριλαμβανομένης της μείωση της εξάρτησης από το πετρέλαιο κλπ. Μέχρι την γραμμή παρελθόν 16 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα τώρα, υπέρ, κατά, ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 23 υπέρ, 25 κατά. Απορρίπτεται. Το δεύτερο τμήμα. Τρίτο τμήμα. Από τη λέξη roads. Η λέξη road μάλλον. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική ε. Καθορισμός εξωτερικού κόστους. Και δώσε τμήματα. Πρώτον, το σύνολο με εξαίρεση συμπεριλαμβανομένου της μείωσης της εξάρτησης από το πετρέλαιο και ρόλι. Πέρα. Κατά αποχές εγκρίνεται το πρώτο τμήμα. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος. σοσιαλιστική ψήφο επιπλέον. Σηκώστε, βγάλε την κάρτα σας. Πέρας. 23 υπέρ, 25 κατά. Απορρίπτεται όπως και πριν. Τρίτο τμήμα, Roads υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική F, σίγμα ΑΦ Και εδώ χωριστή ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα, όλος ο συμβασμός χωρίς τη λέξη road. Και λογή κλίματος. Όχι, είναι όλος ο συμβασμός με εξαίρεση τη λέξη road. 2012 στη δεύτερη παράγραφο, αλλαγή κλίματος στην παράγραφο 2, στην παράγραφο 2 της 2 not και το πρώτο και δεύτερο τμήμα στην παράγραφο 2 β. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα η λέξη road υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τρίτο τμήμα 2012 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τέταρτο τμήμα climate change υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται πέμπτο τμήμα παράγραφος 2.2 υπέρ κατά ηλεκτρονικός έλεγχος στο πέμπτο τμήμα. Εδώ έχουμε έναν του ΕΛΚ επιπλέον. Πέρας. 24 υπέρ, 23 κατά. Καμία αποχή εγκρίνεται. Έκτο τμήμα. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Έβδομο τμήμα. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία του συνδέφου Λίχτεμπεργκερ που προστίθεται στην ε, συμβαστική σίγματα. Προσθέτεται η λέξη effectiveness όπως αναφέρεται στο παράτημα 3 για να γίνει πιο αποτελεσματικό. Ποιες είναι υπέρ της προφορικής Λίχτενμπέργκερ. Κατά αποχές δεν εγκρίνεται. Δεύτερη προφορική τροπολογία Λίχτενμπέργκερ. Η έκθεση θα πρέπει να συνδέεται από εκτίμαση των επιπτώσεων που θα έχει κλπ. λοιπά Υπέρ, κατά, εποχές απορρίζονται και αυτή. Ηλεκτρονικός έλεγχος, ηλεκτρονικός έλεγχος. Στην δεύτερη προφορική τροπολογία Λίχτεμπεργκερ. Hanno votato tutti, Ψηφίσατε όλοι πέρας. Έχουμε 18 υπέρ, 29 κατά. Μία αποχή απορρίπτεται. Συμβαστική ε, G, Z, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. H, Ι, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. E, Θ, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 160 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 161 de Grand Pasquale υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 162 Αγιάλα Σέντερ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 163 υπέρ κατά έλεγχος 163 19 υπέρ, 29 κατά. Απορρίπτεται. 164 Grand Πασκουάλ υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 165 Μέγερ Μάρκοφ υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 166 Σαβαρή υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. compromise, isn't that yes, yes. Ok. Andiamo all'articolo, all'emendamento 12. Itra 12 19. Τροπολογία Ήτρα 19. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Το δεύτερο μέρος του συμβιβασμού ε νομίζω ότι έχει απορριφθεί. Δηλαδή το 11 θεωρείται ότι, έχει, ότι δεν έχει υιοθετηθεί. Με συγχωρείτε. Bene, metto in votazione. Ψηφίζουμε την τροπολογία Ήτρα 20. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 178 κατέπεσε. Και οι υπόλοιπες καταπίπτουν. 198. The Grand Pasquale. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 200. Λίχτενμπεργκερ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 202 Λίχτενμπεργκερ υπέρ κατά αποχές απορρίπτει 203 αποσύρθηκε 204 Λίχτενμπεργκερ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 205 Κώστα Κοτσιλόβο υπέρ κατά Αποχέ απορρίπτει 206 Λάχτφριντ υπέρ κατά αποχές απορρίπτει 207 Γέγκλ υπέρ κατά αποχές απορρίπτει 208 Στόκμαν υπέρ κατά αποχές απορρίπτει 209 Λάχτφριντ υπέρ κατά αποχές απορρίπτει 210 Βατάνεν υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 211 φέρμπερ κατά αποχές απορρίπτεται 212 διγκράμμ πασκουάλ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 213 δεβέρακ Θέλετε τη 212 ηλεκτρονικά. Μάλιστα, 212. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 18 υπέρ 29 κατά. Καμία αποχή απορρίπτεται. 213 αντεβέρακ υπέρ. Κατά. Αποχές. Η κυρία Αντεβερά κέρδισε τη λοτερία σε αυτή την περίπτωση. Συγχαρητήρια. Και τώρα πηγαίνουμε στην 13 του εισηγητή. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ήτρε 22. Ναι, είναι αποδεκτή υπέρ, κατά, ηλεκτρονικός έλεγχος, ήτρε 22. Πέρας, 24-24. Απορρίπτεται. 14 ισχυρή υπέρ κατά ηλεκτρονικός έλεγχος η 14. Πέρας. 25 υπέρ, 22 κατά. Καμία αποχή εγκρίνεται. 220 Βόρτμαν Κόλ, Γερζεμπόφσκι. Ω προσθήκη. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Δεκαπέντε του εισηγητή. 221 για Λασέντε, 222 την Γκραν Πασχόλ Καιρό. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. πέπτη 223. 16 του συγητή υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 225. Ενής Με προφορική τροπολογία της κυρίας Βόρτμαν Κόλ. Σας διαβάζω την παράγραφο. Ε, κόστες στο χρήστη θα είναι ανάλογα με την διάρκεια της χρήσης της υποδομής ή τις η ημέρα, μήνα κλπ. Ιδιαίτερα τη μηνιαίο τέλος δεν θα είναι πάνω από το 10% του ετησίου τέλος. Το εβδομαδιαίο δεν θα είναι πάνω από το 5% του ετησίου και το ημερήσιο συντελεστή δεν θα είναι παραπάνω από 2% από τον ετήσιο συντελεστή. Αυτό προσθέτει η προφορική τροπολογία. Έχετε το λόγο ο εισηγητή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε επειδή το, τη συζητήσαμε την τροπολογία αυτή και και εγώ σκέφτηκα πώς πρέπει να γίνει η διατύπωση. Δεν έχω καμία αντίρρηση να αποδεχθούμε αυτή <clears throat> τη διατύπωση, αλλά νομίζω ότι άργησε πάρα πολύ να υποβληθεί. Και γι' αυτό ο συντάκτης της αρχικής τροπολογίας δεν συμφωνεί με αυτή τη ε, διατύπωση ε, προτείνω λοιπόν να την απορρίψουμε και να προσπαθήσουμε να βρούμε μια καλύτερη λύση μέχρι την Ολομέλεια. Δηλαδή νομίζω ότι αυτή τη στιγμή θα έπρεπε μάλλον να το απορρίψουμε αλλά εσείς θα λάβετε την τελική απόφαση. Μπορείτε να ψηφίσετε την τροπολογία. Εγώ όμως σας προτείνω να μην τη στηρίξουμε τώρα, αλλά να την προωθήσουμε στην Ολομέλεια και να την ξαναδούμε εκεί. Δηλαδή δεν έχετε αντίρρηση να ψηφίσουμε την τροπολογία, εσείς όμως προτείνετε ότι ασχέτως του αποτελέσματος το πρόβλημα αυτό θα πρέπει να το ξανασκεφτούμε ε, και να δούμε τι θα γίνει στην Ολομέλεια. Οπότε υποβάλλω προς ψήφιση την τροπολογία Hens-Jensen όπως έχει ε, τροποποιηθεί από την τροπολογια wortmann Wortman-Koll, ο κύριος Στέρξ. Κύριε ε, Πρόεδρε, οι συντάκτες της ε, αρχικής τροπολογίας δεν, ε, έχουν, δεν επιμένουν να διατηρηθεί η αρχική τροπολογία. Θέλω δηλαδή να συμφωνήσω με τον συνάδελφο και μπορούμε ενδεχομένως στην Ολομέλεια να διερευνήσουμε μια άλλη λύση. Μπορούμε το να ψηφίσουμε. Εντάξει, θα βρούμε μία λύση, αλλά είναι ένα πολύ βασικό θέμα και έτσι πρέπει να βρούμε μία λύση. Πρόεδρος, θα ψηφίσουμε την τρολογία Χένης Πασκάρτ ως έχει αρχική μορφή και λαμβάνουμε υπόψη του τι υπόθηκε εδώ και τι δυνατότητα υπάρχει για παρέμβαση για να ληφθεί υπόψη και η πρόταση Βόρκμαν Κόλ μετά την ψηφοφορία. Ψηφίζουμε την 225 χωρίς προφορική τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Ένις Πρασκάρ Γιένσεν. Έχουμε έναν του ΕΛΚ επιπλέον. There is an extra PPA. E. Ok. Chiusa la votazione. Πέρας. 28 υπέρ, 17 κατά. Εγκρίνεται. 17 του εισηγητή. Ταυτόσιμο με την Αγιάλα Σέντερ 228, Φέμπε 229, 230 Γκραμ Πασκάλ, 231 Βατάνη και Ήτρα 22. Υπέρ. Σχεδόν όλοι. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Ήτρε 24 υπέρ κατά αποχές απορρίβεται. ...232 Φέρμπερ και 233 αποσύρθηκε 232 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτε 2.34 life free repair κατά αποχές εγκρίνεται ηλεκτρονικός έλεγχος τη 234 Ψηφίσατε όλοι. Και πάλι έχουμε έναν ΕΛΚ παραπάνω. Λίγη ψηφοφορία. 25 υπέρ, 23 κατά, άρα εγκρίνεται. Και τώρα προχωράμε στην 252 ε, σημείο, άρθρο 1 σημείο 2 η τροπολογία Wortman Collar για Ζεμπόρσκι υπέρ. Κατά. Αποχές νομίζω ότι απερίφθη, αλλά είμαστε πολύ τσιματσίμα, οπότε ας ξεκινήσουμε για τον έλεγχο ηλεκτρονικά της 252 Βόρτμαν Κόλ για Ψηφίσατε όλοι. Λίγη ψηφοφορία. 22 υπέρ, 26 κατά, απορρίπτεται. Πάμε στη 253 Φεράρι, υπέρ. Κατά. Αποχές, απορρίπτεται. 200 262 Αλμπερτίνη Γαβρόνση Ντεγκάντη Πρασκουάλ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 19 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 265 ρακ υπέρ κατά αποχές και αυτή απορρίπτεται. ...264 Λίχτενμπέργκερ... ...που είναι η ίδια με την Ήτρεβε 26... ...υπέρ... ...κατά... ...αποχές... ...απορρίπτεται... ...πάμε στη 266... Φεράρι. Το πρώτο μέρος, διότι το δεύτερο κατέπεσε εφόσον υπερίσχυσε ο συμβιβασμός 1. Λοιπόν, είναι... λοιπόν μόνο το πρώτο μέρος, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 268 αδεγιάλα σέντερς, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 270 Αλμπετίνη Γκαβρόνσκι που είναι ταυτόσιμη με τη 271 Φεράρι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για αυτά. Ξεκινά ο έλεγχος. 270 Αλμπερτίνη Γκαβρόνσκι και Γκραντε Πασχουάλ και Φεράρι που είναι ταυτόσημη. Ψηφίσατε όλοι. Κλείνει η ψηφοφορία. 19 υπέρ 26 κατά, άρα δεν εγκρίνεται. Και προχωρούμε στην 272 Στόκμαν υπέρ. Κατά, αποχές εγκρίνεται. Και αυτό οδηγεί στην κατάρριξη της 273, πάμε στη 274 υπέρ, κατά, αποχές Απορρίπτεται. 275. Γκρός. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 275 καταπίπτει. 277 γκρός. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται και άρα καταπίπτει 278. 279 Μέγερ Μάρκοφ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 280 Μέγερ Μάρκοφ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 281 Ντεγκράντε Πασχουάλ Γένσεν που είναι το ταυτόσιμο 282 Γέγκλ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 283 Λάχτριντ, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 284 ρακ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 20 του εισηγητή που είναι ταυτόσιμη με τη 285 Lightfried και 286 Μέγερ Μάρκοφ υπέρ κατά Νομίζω ότι εγκρίθηκε, αλλά κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο, ξεκινά. Ψηφίσατε όλοι. Λίγη ψηφοφορία. Ψήφισαν 46. 24 υπέρ, 22 κατά, άρα εγκρίνεται. Πάμε στη 287, Λάιχτφριντ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τώρα ψηφίζεται 288. Αλμπερτίν Καβρό Ιδεράρη υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Θέλετε να ελέγξουμε ηλεκτρονικά, ελέγχουμε. Ξεκινάει η ψηφοφορία για τη 288. Ψηφίσατε όλοι. Ναι. Λίγη ψηφοφορία. 25 υπέρ, 21 κατά, άρα εγκρίνεται. 289 καταπίπτει και πάμε στη 290 λάιχτριτ. Ποιο είναι υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. The Grand Pasquale, 291 καιρό. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 292. Λάιχτφριντ υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 293. Ε, Ένις Πλασκάρου Διάννησεν υπέρ. Κατά. ΦΕΣ απορρίπτεται. 294 Λάιχτφριντ. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 295 Λάιχτφριντ. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 296 ΛΑΙΧΤΡΙΤ, Ταυτόσημη με τη 297 Blockland 298 Γιάκοψ. Υπέρ. Κατά. Και αυτή νομίζω ότι απερίφθη, ας κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο γιατί ίσως κάποιος ε, δεν σήκωσε το χέρι του. Ε, γιατί 296, 97, 98 ψηφίσατε, δεν υπάρχουν ε, πλεονάζοντες, υπάρχουν πάλι πλεονάζοντες ΕΛΚ. Κύριε Γιατζεμπόσχη, για φροντίστε το. Τώρα είμαστε εντάξει. Λίγοι. 22 υπέρ, 25 κατά, μία αποχή, άρα απορρίπτεται. Και πάμε στη 299 μπάρση πατάκι που είναι ταυτόσιμη με την Ήτρε 27. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Μπλόκλαντ 300 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται αποσύρεται η 301, η 302 μπαρ στη πατάκι έχει καταπέσει διότι υπερψηφίσαμε 300 και πάμε στην 303 Λάχτφριντ, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Οι 304 και 5 είναι ταυτόσιμες ποιες είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 306 Λάχτφριντ υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 307 Λάχτφριντ υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τώρα, οι άλλες έχουν καταπέσει και πάμε στην 310 Φεράρι, υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. 311 Λάιχτφριντ, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 312 Βατάνερ, υπέρ κατά, αποχές, νομίζω ότι εγκρίθηκε, ας ελέγξουμε. Την 312 βατάνεν. Ψηφίσατε όλοι, 48 ε, ψήφισαν, 25 υπέρ, 22 κατά, άρα εγκρίνεται. 313 Λάιχτριντ υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 319 ε, Γκράντες Pascual και υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 314 Γκουρμάι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 315 Φέρμπερ υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 318 Λοκούρτου Πατριτσέλο Ζαπαλά υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 316 Αλμπερτίνη και Ρώση Φεράρι ε, και η, η ταυτόσημη με την Φεράρι 317 αλλά εδώ λέει όχι εντάξει είμαστε άρα ψηφίζουμε 316 και 317 ποιος είναι υπέρ κατά Αποχές νομίζω ότι απερίφθη ηλεκτρονικός έλεγχος γιατί είναι κάπως ασαφές. Ψηφίσατε όλοι. Αν ψηφίσατε όλοι, ψηφίσαν 45, λίγη η ψηφοφορία, 14, 17 υπέρ, 28 Κατά δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. 320 Λοκόρτο πριτσέλο Ζαπαλά. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 321 Λίχτενμπέργκερ. Ταυτόσημη με 322 γκουρμά υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 324 Λίχτεμπέργκερ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 325 Λίχτενμπέργκερ ταυτόσημη με την 326 Γκουρμά υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 327 δεκαν, Γκράντες Πασχουάλ Κιερό ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Θέλετε να ελέγξουμε την 327 Ελέγχουμε ηλεκτρονικά 327. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι λίγοι. 22 υπέρ, 26 κατά, απορρίπτεται. 328 γέγκλε, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 329, Λάιχτφριντ, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 330 γκουρμά, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 331 κράντες Πασκάλ καιρό. ποιος είναι υπέρ κατά ε, ε, ξεκινά ο έλεγχος για την 331 ε, κράντες Πασκάλ Κιερό Λίγη ψηφοφορία, 26 υπέρ, 22 κατά, άρα εγκρίνεται. 332 με συγχωρείτε, κατέπεσε τη τροπολογία Παναγιωτοπούλου Κασότου, άρα έχουμε 333 Γιάλα Σέντερ και 334 την Πασκουάλ Κιέρο, ποιος είναι υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι εγκρίθηκε. 335 Γιάλα Σέντερ, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 336 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. «344 μπάτσι πατάκι». Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 345 ρόταν κολ. Ποιος είναι υπέρ. κατά αποχές εγκρίνεται 346 Φέρμπερ που είναι ταυτόσιμη με 347 Γέγκλη υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 348 Μπλόκλαντ υπέρ κατά Νομίζω ότι απερίφθειες κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο στην 348. Ψηφίσατε όλοι. 20 υπέρ, 27 κατά, απορρίπτεται. Η 350, Ένις Πασκάλ Γένσεν. Υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται. 349, Ιβανς. Υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται. 353, Βόρτμαν Κόλ. Υπέρ, κατά. Απορρίπτεται. 351 Λάιχφιλντ, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 352 Λίχτενμπεργκερ υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 22 του εισηγητού υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 354 Χένις Πασκαριένσερ υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 3.55 ελάχιστο. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Και Καταπίπτουν κάποιες ενδιάμεσες, φτάνουμε στην 364. Υπέρ, κατά, αποχές, Απορρίπτεται. 365. Περ, κατά, αποχές, γκρίνεται. 376 σουτ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 377 Wortman Collier Ζεμπόσκι. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 378 Στέρξ. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ακόμη και ο κύριος Στέρξ μπορεί να έχει κάποια στιγμή επιτυχίες. 23, ραπορτέρ, ε, εισηγητού, υπέρ, κατά, αποχές. Όχι, αυτό καταπίπτει. 371. 372. που είναι ταυτόσιμη με την 373. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συγγνώμη για τον κύριο Σαβαρή. 385. Γέγκλ. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 24 του εισηγητού υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Andiamo al 25 del relatore. 25 του εισηγητή ως προσθήκη στο συμβασμό F τροπολογία στο άρθρο 1, 6 το άρθρο 11 παράγραφος 1 και 1α νέο υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 394 λαιχτφριντ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ερχόμαστε στο άρθρο 2, 2.24-2.25 υπέρ Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι πρέπει να ψηφίσουμε την 4.23 ως προσθήκη. Μάλιστα, έχετε δίκιο, λέει ο Πρόεδρος, ως προσθήκη στον συμβαστική F σίγματα αυτές, 23 λοιπόν, υπέρ, κατά, αποχές αυτό εγκρίθηκε όχι θέλετε ηλεκτρονικό έλεγχο ναι εγκρίθηκε χάρη στην κυρία Βόρτμαν Κόλ ερχόμαστε στο 424 την Πάσκολα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 424-425 428 Lightfield υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 33 ηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 34 ηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 35 ηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τετρακόσια πενήντα ενίς υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 458 για Σέντερ υπέρ. Κατά αποχές απορρίφεται. 459 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 460 Λίχτεμπεργκερ υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 94 στο άνεξ στο παράρτημα τετρακόσα ογδόντα οχτώ Βόρτμαν Κόρια Ζεμπόφσκι 488 υπέρ κατά αποχές αποχές 489 Ένις πλασκαρι υπέρ κατά αποχές απορρίβεται 490 light thread υπέρ κατά αποχές απορρίβεται 491 Jacobs υπέρ κατά αποχές απορρίβεται 493 Λάιχφριντ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 494 495 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 496 Lightfried υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 498 Ένις Πλασκάρτη Γένσεν υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος 498 πέρας 23 υπέρ 25 κατά απορρίπτεται 24 υπέρ 25 κατά απορρίπτεται 499 Jacobs υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 500 Evans υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 501 Evans υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 502 κόρ για Ζεμπόφσκι ταυτόσιμη με την 503 Ενίς Πλασκάρ υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 504 λάχθη διπέρ. κατά αποχές απορρίπτονται 505 λάχθη διπέρ. κατά αποχές απορρίπτονται 506 Βότμαν Κόλ Γένσεν καταπίπτει Κατά καταπίπτει μέχρι και την 514. 515 λάχιστον υπέρ κατά αποχές απορρίπτει. 516 λάχιστον υπέρ κατά αποχές απορρίπτει. 517 λάχιστον υπέρ κατά αποχές απορρίπτει. Όχι 518. 5.19 είναι σπλασκάλτς και 5.20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 529 Εύανς υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 39 συγητής υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 522 έβανση υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 40 συγητής υπέρ κατά απόχέ απορρίπτεται 523 Ένις Πασκαρι Πέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος 523 Πέρας 21 υπέρ 25 κατά απορρίπτεται 529 Λάιχτφριντ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 530 όχι 42 The Grand Pasquale υπέρ ναι έχετε το λόγο Θα ήθελα να μου πείτε πριν να περάσουμε στην ατολική σκέψη το παράρτημα τροπολογίες 500. 12, 13 και 14 δεν τις ψηφίσαμε. Δεν καταλαβαίνω όμω για ποιο λογο ah, ah, uh, Στην κατάλληλη ψηφοφοριών φαίνεται ότι καταπίπτουν διότι στην τελευταία εκδοχή που είχε το γραμματείο, η γραμματεία δεν εμφανίζεται. Οι 512 και οι 513 δεν ψηφίστηκαν διότι καταπίπτουν. Ιδεολογικές σκέψεις λοιπόν. η Πασχουά καιρό 42 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Τι κάπως ήρθηκε. Οι άλλες καταπίπτουν από 44 47. Ήτρε 1. Υπέρ κατά εγκρίνεται 49 Λάιφριντ πέρα. κατά αποχές απορρίπτε 50 Ρακ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 51 Παναγιωτοπούλου υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ήτρε 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτε ή 3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτε 52 τικάου με ήτρε 4 υπέρ κατά αποχές απορρίπτε εισηγητής αριθμών 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται καταπίπτουν 53, 54, 55, 56, 57, Ερχόμαστε στη τροπολογία 2 του εισηγητή. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 3 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 60 Βόρτμαν Κόρια Ζεμπόφσκι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 4 του εισηγητή κατέπεσε αιτιολογική σκέψη 7 66 στέρεξη υπέρ 66 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 67 καταπίπτει. 68 Λίχτεμπεργκερ. υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτει. 5 του εισηγητή υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται από 69 καταπίπτουν 71 ελάχιστον υπέρ καταπίπτει και αυτή υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 6 του εισηγητή συμβατή με τη συμβαστική α υπέρ Υπαριθμών 6 του εισηγητή. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 78 Στόκμαν υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 79 λάχιστον. υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Ήτρα 6. υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 80 ελάχιστον υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται καταπίπτουν 81, 7, 82, 83 στόκμαν υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 103 κατέπεσε εν μέρη. Ένα τμήμα μέρη ψηφίζουμε. 103 βότμαν Κόλ υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 109 βότμαν Κόλ υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 110 Κώστα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 111 καταπίπτει 112 likes υπέρ κατά αποχές Η 20 εγκρίθηκε, άπρεπε να ψηφίσουμε την 113 ΡΑΚ, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. καταπέπτουν από 114. Πάμε στην 119 Lightstream υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 120 Φέρμπερ, 121 και 122 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 123 Δεγκράμ Πασκουάλ υπέρ κατά αποχές απορρίπτει 124 γκρός υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ήτρε 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτει 125 κόστα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 126 στέριξη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 127 βαρμαν Κόλια Ζεμπόφσκι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 143 κατά καταπίπτει 128 γέγγλια υπέρ κατά αποχές απορρίπτει 129 Φέρμπερς 130 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτει 100 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ήτρ 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Εκατόν σαράντα ένα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 150. Λίχτενμπέργκερ και Ήτρα 14 επίσης υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 151 Βόρτμαν Κόλ υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 154 Λίχτενμπέργκερ υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Ήτρε 15 υπέρ. Κατά αποχές κατά πίπτη 155 Λίχτενμπεργκερ υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Ήτρε 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 156 γέγκλα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 10 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 157 κατά καταπίπτει 158 Αγιάρα Σέντερ υπέρ κατά αποχές απορρίβεται ήτρε 17 υπέρ κατά αποχές απορρίβεται και ψηφίζουμε το σύνολο της νομοθετικής πρότασης ηλεκτρονικά. Το ΕΛΚ έχει μία επιπλέον ψήφο. Ψηφίσατε. Πέρας, επί 47, 31 υπέρ, 16 κατά. Εγκρίνεται. Και περνάμε στη δεύτερη ψηφοφορία. Τώρα το νομοθετικό ψήφισμα και χειροκροτήστε μετά από αυτό. Τώρα ψηφίζουμε πάλι ηλεκτρονικά. Πάλι έχουμε μία επιπλέον του ΕΛΚ. Πέρας. 46 ψηφίζουν. 32 υπέρ, 14 κατά. Αποχή 0. Πέρας αυτή τη ψηφοφορία. Συγχαρητήρια στον εισηγητή μας και σε όλους όσοι συνεργάστηκαν. Τώρα δεν τελειώσαμε. Υπομονή. Άλλη μία ψήφος και τελειώσαμε. Metto in votazione, per favore, votiamo sul rapporto di iniziativa. Λοιπόν, έχουμε την έκθεση πρωτοβουλία δέσμη οικολογικών μεταφορών και εσωτερήκευση του εξωτερικού κόστου. Greening. Έκθεση για Ρεζεμπόφσκι. Καταρχήν τι συμβαστικέ.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 εγκρίθηκε. Συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. συμβαστική 8 ηλεκτρονικά. πέρος επί 40, 22 υπέρ, 17 κατά εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 10 χωριστά τμήμα. Το πρώτο τμήμα έχει απογοητευτεί από το ότι υπέρ, κατά, ηλεκτρονικός έλεγχος πρώτο τμήμα της συμβαστικής 10. Επί 38, 29 υπέρ, 8 κατά εγκρίθηκε. Το δεύτερο τμήμα το υπόλοιπο υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 11 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνονται. Συμβαστική 12 πρώτο τμήμα, πρώτο notes that the commission as they see fit. Υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα and secondly μέχρι member states discretion. Υπέρ, κατά ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψήφισαν 40, πέρασε. Επί 41, 19 υπέρ, 22 κατά. Άρα το δεύτερο τμήμα δεν εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται το τρίτο. Τελειώσαμε με τις συμβαστικές τροπολογίες. Τώρα να δούμε τι επιζεί. Δέκα τικάου υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τη δέκα. 14 κατά απορρίπτεται. 14 Λίχτενμπέργκερ υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 15 Γιάλα Σέντερ υπέρ. Κατά αποχή εγκρίνεται. 19 σεβαρή υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 33. Τεσενή. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίβεται. 32 Λίχτενμπεργκερ υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 32. Πέρας. 25 υπέρ 17 κατά εγκρίνεται. Τριάντα εννέα. Λίχτεμπεργκερ υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 40 σαβαρή υπέρ κατά αποχές απορρίπτε 41 Λίχτεμπεργκερ υπέρ κατά ηλεκτρονικός έλεγχος 41 Πέρασε. 9 υπέρ 33 κατά. 64 Αγιάλα Σέντερ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 65 Αγιάλα Σέντερ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 71 ένα Λάιφριντ υπέρ κατά αποχές απορρίπτει. 72 αλκαντράβι υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος 72 72 Ελκαντράβη πέρας 24 υπέρ 18 κατά εγκρίνεται 74 Λίχτενμπεργκερ υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 75 Σαβαρή υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 77 Φεράρι. και 78 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Νέα παράγραφος μετά την... 14. Μετά τη 14. 76 σαβαρή. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 1. Σαβαρή. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2. Δεσενέ. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται ηλεκτρονικός έλεγχος 2-9 42 ψηφίζουν. Δεκαοκτώ υπέρ, 24 κατά απορρίπτεται. Τρία Ελκαντράου υπέρ. κατά ηλεκτρονικός έλεγχος στα 3. Πέρασε. Απορρίπτεται με μεγάλη πλειοψηφία. 4 σαβαρή υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 5 σαβαρή υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 6 ελκαντράου υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 8 Λίχτενμπέργκερ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 9 ελκαντράου υπέρ κατά αποχές απορρίπτε Εφτά γέλα σύνδερ υπέρ κατά αποχές απορρίπτε τελική ψήφος Πέρας. Επί 42, 26 υπέρ, 16 κατά. Καμία εποχή. Συγχαρητήρια κύριε Γιαζεμπόφσκι. Εγκρίθηκε και αυτή η έκθεση.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 Alors, on va reprendre nos travaux. Θα συνεχίσουμε τις εργασίες μας. Παρακαλώ να καθίσετε στη θέσεις σας. Περνούμε στο σχέδιο δράση για την αστική κινητικότητα, σημείο 12. Εισηγητής, ο κύριο Σαβαρή, του δίνω μέσω το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας παρουσιάζω την έκθεση αυτή, η οποία είναι κάπως ιδιόμορφη, διότι όπως γνωρίζετε, συμπεριλαμβάνεται στα πλαίσια μιας πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που στην πράξη κατέληξε να πράσινο βιβλίο της 25 Σεπτεμβρίου 2007 και τον Ιούλιο του 2008 κατέληξε μια σημαντική έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με ψήφισμα του συναδέλφου Γάινε Ρακ. Ως συνήθως, τα πράσινα βιβλία σε επίπεδο κομίσιο έχουν ως στόχο να συμπεριλάβουν απόψεις ενδιαφερομένων οργανώσεων και πολιτών το θέμα αυτό και καταλήγουν σε ένα σχέδιο δράσης το οποίο μας αναγγέλλεται. Καταρχάς το σχέδιο αυτό είχε τεθεί σε κίνηση από τον Επίτροπο και πολλές φορές είχαμε πει ότι θα πρέπει σε θέματα αστικής κινητικότητας να παρέμβουμε. Τι συμβαίνει τώρα. Το σχέδιο δράσης το οποίο είχε αναγγελθεί για το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο όλο και περισσότερο αναβαλόταν και καθορίστηκε η ημερομηνία καταληκτική της 10ης Δεκεμβρίου και ο Επίτροπος Ταγιάννη με πολύ τάκτ, διότι εγώ πρέπει να σας πω ότι ορίστηκα εισηγητής του σχεδίου δράσης, με ενημέρωσε ότι είχε κάποιες δυσκολίες και θα προσπαθούσαν το δημοσιεύσει στις αρχές του Ιανουαρίου. Αποφασίσαμε λοιπόν, και σας λέω αυτό είναι το ιδιόμορφο στοιχείο, να παρακάμψουμε το σχέδιο δράσης της Επιτροπής και να το επομιστούμε. Τι να κάνουμε. Ένα σχέδιο πρωτοβουλίας. Ένα ως κοινοβούλιο προτείνουμε εμείς στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή ένα σχέδιο δράση για την εθνική κινητικότητα χωρίς να είμαστε, αρμόδιοι τελικά. Δεν είναι όμως η μόνη ιδιομορφία αυτής της υπόθεσης, δεδομένου ότι δεν έχουμε ακόμη τα αποτελέσματα του πράσινου βιβλίου και της διαβούλευσης της Κομισιόν, τα οποία τα έχει κλειδωμένα σε ένα σιρτάρι. Κρυφά η Κομισιόν προς το παρόν. Χρειάστηκε λοιπόν, χωρίς να έχουμε στη διάθεσή μας αυτά τα στοιχεία της αρχικής διαβούλευσης να προχωρήσουμε, για να προτείνουμε το δικό μας σχέδιο δράσης. Ποιος είναι ο στόχος αυτού του εγχειρήματο. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω το σύνολο των πολιτικών ομάδων, δεδομένου ότι είναι ασύνηθε το θέμα αυτό και θα ήθελα θέλω να ευχαριστήσω τον Ράιν Ρακ, δεδομένου ότι το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του είχε αποφανθεί για την Πράσινη Βίβλο. Ο στόχος αυτού του εγχειρήματο είναι πρώτα απ' όλα να διαμαρτυρηθούμε για τη στάση αυτή της Επιτροπής σε σχέση με τις δεσμεύσεις που αναλάβει καταρχάς και πρέπει να πω ότι ενισχύθηκε αυτή η πρωτοβουλία μας για την ε, πρωτοβουλία των στη επίσημη συζήτηση τον Ιανουάριο που κάναμε με την Κομισιό θέσαμε το σχετικό ερώτημα και είδαμε ότι υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον εκ μέρους της Επιτροπής ίσως με διαφορετικές χωριστές πρωτοβουλίες, αλλά χωρίς να καταλήγουν όλα αυτά σε ένα εγγύς τουλάχιστον και συγκεκριμένο μέλλον σε πρωτοβουλία. Γι' αυτό θελήσαμε εμείς να υποβάλουμε τις πιο λειτουργικές, συγκεκριμένες και πρακτικές ερωτήσεις, ώστε παρά τη γνώση ότι δεν θα έχει νομική αξία δικό μας οχήρημα, να οθήσουμε στην Κομισιόν στο να κάνει κάτι στον τομέα αυτό. Γιατί πιστεύουμε ότι αυτό είναι αναγκαίο. Πρώτα απ' όλα, διότι όπως γνωρίζετε οι μεταφορές είναι αρμοδιότητα κοινή μεταξύ κρατών μελών και ευρωπαϊκών κοινοτήτων μία από τις πιο σημαντικές δραστηριότητες σε θέματα συναπόφασης. Και δεν μπορούμε οι αστικές συγκοινωνίες να είναι ένα θέμα το οποίο θα παραγνωρίσουμε, διότι 60% των πολιτών ζουν σε αστικές περιοχές, το 2020 το 80% θα έχει, σε 80% θα έχει ανέβει αυτό το ποσοστό. Άρα οι αστικές συγκοινωνίες, όπως καταλαβαίνετε, είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό και δεν μπορούμε να αγνωρίσουμε εμείς ένα γεγονός τόσο μεγάλης εμβέλειας. Δεύτερος λόγος ψηφίσαμε το πακέτο για το κλίμα τον Δεκέμβριο και κατά ελληνικό τρόπο τη στιγμή κατά την οποία οι αρχικές των κυβερνήσεων χαιρετίζουν το πακέτο για το κλίμα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πράττει το ίδιο, μας αναφέρουν το οποιαδήποτε σχέδιο δράσης για τον τομέα αυτό των ε, αστικών μεταφορών. Ξέρετε πόσο σημαντική είναι και η συμβολή του για τη διαμόρφωση του κλίματος και για τη χειροτέρευση του κλίματος. Η είναι οι μεταφορέ υπεύθυνε 70%. Άρα θα πρέπει να ενεργήσουμε. Πώ θα ενεργήσουμε, Πρόκειται για ένα ευαίσθητο θέμα, διότι η οργάνωση των αστικών συγκοινωνιών τη αστική κινητότητα είναι κάτι το οποίο είναι στα στην αρμοδιότητα και στα χέρια της τοπικής αυτοδιοίκηση των τοπικών αρχών και βεβαίως δεν μπορούμε εμείς να μην συμβαστούμε την ε, κυρίαρχο εξουσία αυτών των ε, διοικήσεων τοπικών και δεν μπορούμε σε αυτό το επίπεδο να επιβάλλουμε το οτιδήποτε σε οποιαδήποτε επίπεδο. Δεδομένου ότι ένας γενικός κανόνας θα είναι ούτως ή άλλως αντίθετος στην αρχή της επικουρικότητας και βεβαίως δεν θα λαμβάνει υπόψη την πολυπλοκότητα και την ε, ποικιλομορφία των διαφόρων καταθέτων. Η πρώτη λοιπόν αρχή είναι απόλυτος σεβασμός της αρχής της επικουρικότητας. Αντιθέτως όμως θεωρούμε ότι όπως σε πολλούς τομείς η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να είναι μία υπεραξία. Πρώτα απ' όλα, για να υπάρχει καλύτερη ενημέρωση και να γνωρίζει κανείς καλύτερη πραγματικότητα των αστικών μεταφορών που στατιστικά σήμερα δεν είναι γνώστα σωστή, να διευκολυνθεί η ανταλλαγή των πρακτικών να μπορέσουν τα δίκτυα των διαφόρων πόλεων και οι διάφοροι οργανισμοί υπεύθυνοι για τις ε, ε, μεταφορές να βρίσκονται σε συνεχή διάλογο. Άρα το πρώτο σκέλος αυτό είναι πολύ σημαντικό και αφορά όλα αυτά τα οποία σας προανέφερα, την δημιουργία δικτυακής πύλης για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, στοιχείων, μόνιμο φόρουμ των ε, υπεύθυνων οργανισμών αστικών συγκοινωνιών για την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών, βελτίωση των τα με την ε, σύνδρομη της Eurostat και εδώ σας λέγω ότι δεν θέλουμε όπως γίνεται αυτομάτως να κάνουμε ένα νέο ευρωπαϊκό οργανισμό ο οποίος να ασχολείται με το θέμα αυτό. Έχουμε τα απαραίτητα όργανα σε όλα τα επίπεδα για να ασχοληθούν με τα θέματα αυτά ενίσχυση του προγράμματος Σίβητας που μέχρι σήμερα ήταν το μοναδικό σημαντικό μέσο μας επέντευξη να κάνουμε την ανταλλαγή βελτίστων πρακτικών και να κάνει ε, μειωτικούς διαγωνισμούς για πολύ καινοτόμα σχέδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω αυτού του μέσου, αλλά θα θέλαμε επίσης και για λόγους διαφήμισης και για την διαπαιδαγώγηση της κοινή γνώμη να έχουμε και ένα βραβείο το οποίο θα απονέμεται την ημέρα της εθνής κοινοτικότητας και θα αφορά το σύνολο όλων των αστικών περιοχών. Γι' αυτό λοιπόν θέλουμε να κατανοήσουν καλύτερα και με πιο διαφανή τρόπο όλοι περί τίνος πρόκειται να ανεμηθούν καλύτερα. Δεύτερο, βελτιστοποίηση των διαφόρων τρόπων μετακινήσεων με καλύτερη και προγραμματισμένη ενημέρωση. Και δεν θέλω να πω ότι θέλουμε να πούμε ότι κάποιος προτιμά το αυτοκίνητο από το σιδηρόδρομο ή όχι. Θέλουμε να δούμε πώς θα κάνει την καλύτερη αξιολόγηση των συστημάτων μετακίνησης, που είναι πολύ πολύπλοκα, δεδομένου ότι είναι ελέγχοντα μεταξύ τους και σε αυτά τα συστήματα ο κάθε τρόπος μεταφοράς θα έχει το λόγο του, βεβαίως. Τα ιδιωτικά οχήματα, βεβαίως τις συλλογικέ δημόσιες μεταφορές, αλλά και οι ποιες μορφές μετακίνησης που μπορούν ε, να είναι πεζόδρομοι, ε, ειδικοί διάδρομοι για ε, ποδήλατα και ισορροπία στο πλαίσιο των διαφόρων τρόπων μεταφορών. Η πρόταση λοιπόν, η πιο σημαντική στα πλαίσια της έκθεσης είναι ότι θα πρέπει να έχει η Ευρώπη μία προσέγγιση που να δημιουργεί κίνητρα. κίνητρα. Δεν θέλουμε να κάνουμε μόνο περιγραφή του υπάρχοντος συστήματος, αλλά να δημιουργεί κίνητρα. Το κάνει αυτό και σε άλλους τομείς και για τα διαρθρωτικά ταμεία όπου υπάρχουν διάφορες ρυθμίσεις και για την ΚΑΠ που δημιουργεί κίνητρο ώστε να κατευθυνθεί ο Γεωργός στην Α ή Β ε, κατεύθυνση πρέπει να δημιουργήσουμε κίνητρα. Και για να δημιουργήσουμε τα σωστά κίνητρα πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τις αστικές ε, μετακινήσεις και συγκοινωνίες. είτε που θα μοιάζει με το Urban, είτε θα είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θα έχει προσαρμοστεί στις ανάγκες, λαμβάνοντας υπόψη τώρα τους στόχους για την βελτίωση του, ε, των κλιματικών συνθήκων στα πλαίσια των νέων δημοσιονομικών ε, πρακτικών ή θα πρόκειται για ένα ε, διακρατικό πρόγραμμα, αν θέλετε, ούτως ή άλλως είμαστε ακόμη ανοιχτοί. Ο στόχος είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μπορεί εν μέρη να χρηματοδοτεί μελέτες για τα ε, σχέδια αστικών μετακινήσεων και της αστικής κινητικότητας για ε, πόλεις μεγαλύτερων των 100.000 καθήκων, όπου θα λαμβάνεται υπόψη και το φρέτ και η υποστήριξη που χρειάζεται και διπονομής για να γίνει κάτι τέτοιο. Επίσης, όπως στο Urban Transport, λέμε ότι ένα μέρος της χρηματοδότησης, δεδομένου ότι πρόκειται για σχέδιο δράσης και όχι για οδηγία και δεν είναι υποχρεωτικό, ένα μέρος των επενδύσεων να γίνουν με κοινοτική χρηματοδότηση ώστε να έχουμε ένα μόνιμο φόρουμ των υπευθύνων αυτών των αστικών μετακινήσεων, ώστε να γίνεται ενημέρωση για τις καλύτερες πρακτικές, ανταλλαγή εμπειριών. Ζητούμε την Επιτροπή να λάβει υπόψη μελέτες για θέματα τιμολόγησης και ενημέρωσης των χρηστών. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνουν ελκυστικά τα μέσα μεταφορές, ώστε να προσελκυστεί ο χρήστη, να διευκολυνθεί και η ζωή του χρήστη και νομίζω ότι με τις νέες τεχνολογίες και η ενημέρωση είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει πολύ πιο εύκολα. Τρίτος μεγάλος άξονας της πλαίσια τη πρωτοβουλία μα. Έρευνα. Με την βελτίωση ε, των ε, τεχνολογιών, ασφάλεια, εργονομικές κατασκευές, μείωση του θορύβου, διαλειτουργικότητα των μέσων μεταφοράς, όλο αυτό υπέρ του χρήστη. Θέλουμε να υπάρχουν ελάχιστες προδιαγραφές ποιότητας των προσφερωμένων υπηρεσιών για τον χρήστη, κυρίως στα πλαίσια τι οδηγίε για την παροχή καθολική υπηρεσία. Και στο τέλο υποδεικνύουμε, και αυτό είναι κάτι το οποίο θέλουμε να γίνει αμέσω, οι αστικέ συγκοινωνίε να συμπεριληφθούν στο σχέδιο οικονομική ανασυγκρότηση και αναθέρμανση τη Ευρώπη. Γιατί, διότι παντού στην Ευρώπη πρέπει να πω ότι υπάρχουν διάφορα σχέδια τα οποία κρεμούν και μπορούν αμέσω να ολοκληρωθούν. Και τελειώνοντα, ζητούμε από την Επιτροπή να κάνει κάποιες συμπληρωματικές μελέτες και ενδεχομένω να μας δώσει τις κατευθυντήριες γραμμές για κάποιες συγκεκριμένες εμπειρίες τις οποίες θα θέλαμε να αναλύσουμε και να μετρήσουμε. Ζητούμε έκθεση Επιτροπής για τα ιδιώδια στις αστικές περιοχές της πόλης για να δούμε τι γίνεται σε κάποιες πόρες και ποια είναι τα αποτελέσματα, να δούμε αν θα πρέπει να πλαισιωθούν τέτοιου είδους πρωτοβουλίες με γενικές κατευθυντήριες. Πιστεύουμε ότι επίσης θα πρέπει να θεσπιστεί, να δημιουργηθεί ένα δίκτυο πώληση ε, εισιτηρίων για τις αστικές μεταφορές ε, σε σιδηροδρόμους και σταθμούς, ώστε να μπορεί κανείς ε, να αγοράζει με μεγάλη ευκολία τα εισιτήρια του. Δηλαδή, από το Παρί... στο Παρίσι, στην Καρδουινόρ, θα πρέπει κανείς να μπορεί να αγοράσει εισιτήρια για το μετρό του Λονδίνου. Το ίδιο τα αεροδρόμια. Επίσης θα θέλαμε να δημιουργηθεί μια χάρτα των χρηστών και λαμβάνουμε υπόψη και τους ε, ποδηλάτες και τους πεζούς που μοιράζονται όλοι τα ίδια δίκτυα. Και βεβαίω ζητούμε να προωθηθούν και οι ευρωπαϊκές ημέρες χωρίς αυτοκίνητο και τέτοιου είδους παρεμφερείς πρωτοβουλίες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους με των πολιτικών ομάδων οι σκιώδεις ηγητές που με βοήθησαν να συντάξω την έκθεσή μου. Δεν είναι μια έκθεση δική μου, είναι συλλογική και είπαμε ότι πρόκειται για μια πάρα πολύ ε, ιδιόμορφη, έκτακτη ε, πρωτοβουλία την οποία πήραμε και όλη αυτή η διαδικασία μπορούσε να ληφθεί με την πρόσφορα και την συνδρομή όλων των συναδέλφων. Ε, από τη στιγμή την οποία παίρνει μια πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σαν τομέα που είναι αρμοδιότητα, σαν τομέα τη Επιτροπή, πιστεύω ότι καλύτερα να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι τόσο συνενετικό ώστε να είμαστε αποδοτικοί. Βεβαίω αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να κατατεθούν τροπολογίε, αλλά προσπαθήσαμε όλοι εκ των προτέρων να καταλήξουμε σε συμφωνή και σε συνέντε. Θα ευχαριστώ λοιπόν όλου του συναδέλφου και πρέπει να σα πω ότι αυτή η πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει μεγάλη απήχηση και μας υποστηρίζουν όλοι όσοι περίμεναν εκ μέρους της ε, Επιτροπής κάποια πρωτοβουλία. Τα δίκτυα Eurocities, άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς, διάφορες οργανώσεις, πόλεων, οργαν... οι... αυτοί οι οποίοι κάνουν τον εξοπλισμό για τις αστικές συγκοινωνίες και νομίζω ότι εμείς πήραμε τη σκητάλη την οποία παράτησε στη μέση της διαδρομής η Κομισιόν και σίγουρα κάνουμε κάτι το πολύ πιο φιλόδοξο από ό,τι αρχικά προέβλεπε να μας παρουσιάσει η Επιτροπή. Συγγνώμη μακριγώς, ευχαριστώ που με ακούσατε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον εισηγητή σε γενικές γραμμές μπορώ να συμφωνήσω με αυτά τα οποία μας είπε και δεν υπάρχει έκπληξη γιατί ο κύριος Σαβαρή μας είπε ότι αυτά τα οποία υπέβαλε εδώ τα έχει συντονίσει με τους σκιώδεις εισηγητές κατόπιν πολύ λεπτομερούς συζητήσεως ε, για να προετοιμάσει την ομιλία του. Πιστεύω λοιπόν ότι όλα αυτά είναι πάρα πολύ ε, σκόπιμα για να καταλήξουμε σε μία απόφαση. Καταρχήν θα ήθελα να τονίσω τη σημασία αυτής της διαδικασίας. Δηλαδή, αν δεν αναλάβει υπόψη της ε, σοβαρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή την δυνατότητα πρωτοβουλίας του Κοινοβουλίου, τότε το Κοινοβούλιο θα πρέπει πρέπει να πει ότι είναι ανάγκη να γίνει κάτι εδώ διότι εμείς σεβόμαστε το γεγονός ότι υπάρχουν κράτη-μέλη και ιδίως ένα σημαντικό κράτος μέλους όπου υπήρξαν επιφυλάξεις για όλη τη διαδικασία δηλαδή να ασχοληθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τις κρατικές ε, συγκοινωνίες ε, σεβόμαστε αυτό το επιχείρημα και γι' αυτό ε, από εκεί ξεκινούν και όλες οι σκέψεις μας αλλά η επικουρικότητα ε, εφαρμόζεται καλύτερα εάν διατυπωθεί μία πρόταση η οποία λαμβάνει υπόψη την αρχή την επικουρικότητα και αντί να μην κάνει τίποτα και να αφήσει τον πολίτη ε, να μείνει απομονωμένος για να λύσει τα προβλήματα των συγκοινωνιών στις πόλεις. Δηλαδή, όπου μπορεί να υπάρχει ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, πρέπει να τη χρησιμοποιούμε. Και ο κύριος Σαβαρή εδώ ανέφερε μία ε, σειρά παραδειγμάτων που είπε ε, και τονίζει ότι θέλουμε να σεβαστούμε την επικουρικότητα. Είπε ότι δεν θέλουμε εδώ να προδιαγράψουμε τι θα γίνει σε κάθε τομέα, τα να δημιουργήσουμε κίνητρα για να υπάρξουν δυνατότητες οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν εάν ενδείκνυνται για τις ε, συγκεκριμένες τοπικές συνθήκες. Άρα, σεβασμός για την επικουρικότητα και ε, ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Επίσης, ολοκληρωμένη ιδέα Δηλαδή το πρόγραμμα πρέπει να προβλέπει ε, να μπορούν τα διάφορα σημεία να διαπλέκονται ε, γιατί ε, κατά αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να επιτύχουμε το προσδοκόμενο αποτέλεσμα το οποίο δεν είναι τόσο εύκολο να επιτευχθεί. Θέλω να πω εδώ ότι θέλουμε εδώ να συνδυάσουμε την, ε, την ε, πολιτική συγκοινωνιών με άλλες ε, ε, πολιτικές με άλλα ε, θέματα όπως η έρευνα, η τεχνολογία, δηλαδή πολλά θέματα τα οποία συνδέονται με τη συγκεκριμένη ιδέα και ιδίως ε, θέμα προϋπολογισμού, δημοσιονομικών πόρων που χρειάζονται. Βέβαια η τεχνική και η βιομηχανία πρέπει να ενημερωθούν εγκαίρως και θα ζητήσουμε μετά ε, προτάσεις σύμφωνα με τις οποίες οι διάφορες ε, κοινότητες θα μπορέσουν να επιλύσουν πιο εύκολα τα προβλήματά τους και επίσης θα ήθελα ε, να πω ότι ο κύριος Σαβαρή τόνισε επίσης και το πόσο σημαντικά είναι τα δικαιώματα των ατόμων με ειδικέ ανάγκες. Θα μπορούσαμε εδώ να μακρηγορήσουμε αλλά δεν νομίζω ότι αυτό είναι ο στόχος μας γι' αυτό και πάλι θέλω να συμφωνήσω με την έκκληση του κυρίου Σαβαρή Δηλαδή ζητούμε από τους συναδέλφους αυτή την ε, συνεκτική έκθεση να μπορέσουμε να την αποφασίσουμε κατά τρόπον ώστε να την ε, παραδώσουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την δρομολογήση διότι όλοι έχουμε πολλές θαυμάσιες προτάσεις αλλά μην παραμείνουμε με μία σειρά ε, μπαλονιών με αέρα σκέτο εδώ απλούστατα ας προσπαθήσουμε να διατυπώσουμε τις συλλογικές μας σκέψεις που είναι το αποτέλεσμα μιας συλλογικής συζητήσεως κατά τρόπον ώστε να μπορέσουν να υλοποιηθούν. Γι' αυτό και ελπίζω ότι θα υπάρχει μια σαφής ψηφοφορία καταρχήν στην Επιτροπή και στη συνέχεια στην Ολομέλεια διότι είμαστε πεπισμένοι ότι αυτό το πακέτο δράσης είναι αναγκαίο διότι τα προβλήματα της, ε, ε, των εσωτερικών μεταφορών είναι πολύ σημαντικά και πρέπει να τα λάβουμε υπόψη. Ευχαριστώ κύριο Κράμερ. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή διότι ήταν μια ασυνήθιστη συνεργασία, γι, όμως, γι' αυτό όμως και ε, συνεργαστήκαμε ασυνήθιστα, πολλές προτάσεις έχουν περιληφθεί και τον ευχαριστώ και θα ήθελα επίσης ε, ε, να επαναλάβω ότι δεν είναι δυνατόν να συμπεριφέρεται έτσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς το Κοινοβούλιο. Έπρεπε να μας έχει διατυπώσει ένα πρόγραμμα το οποίο δεν έχει πράξει ακόμη Ελπίζω ότι οι παρόντες αυτή την αίθουσα θα αναφέρουν αυτά τα θέματα στους, στις υπηρεσίες τους διότι ξέρουμε ότι προβλέπουμε μία μείωση των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακος αλλά γνωρίζουμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των εκπομπών στις πόλεις προέρχεται από τις συγκοινωνίες και το 70% των βλαβερών εκπομπών προέρχονται από τις συγκοινωνίες και αν δεν λύσουμε αυτό το πρόβλημα δεν πρέπει πλέον να μιλάμε ε, για προστασία του κλίματος διότι πέρυσι κάναμε μία συζήτηση και όλα αυτά αναβληθήκανε διότι στη Γερμανία τουλάχιστον 90% όπως δηλώνει το Υπουργείο Συγκοινωνιών της Γερμανίας τα αυτοκίνητα, οι διαδρομές στην πόλη είναι μικρότερες από 6 χιλιόμετρα. Δηλαδή βλέπουμε ε, ότι αν αναδιατυπώσουμε την κινητικότητα των πολιτών θα μειώσουμε πολύ εύκολα τις ε, εκπομπές και ε, οι δημόσιες συγκοινωνίες δεν είναι ανάγκες μόνο για, την κινητικότητα αλλά και ε, για την βελτίωση του κλίματος. Πιστεύουμε λοιπόν ότι υπάρχει ένας μοχλός διότι εμείς ασχολούμαστε με τις συγκοινωνίες στις πόλεις διότι υπάρχει επικουρικότητα στη, στο, στη Βάδη Βουρτεμβέργη και σε άλλες περιοχές έχει επέμβει το κράτος και έχει ε, ε, λύσει ορισμένα προβλήματα αλλά θεωρούμε ότι η επικουρικότητα είναι απαραίτητη Έχουμε λοιπόν ε, το μοχλό των οικονομικών και γι' αυτό ε, οι πόλεις ε, πάνω από 100.000 κατοίκους πρέπει να υποβάλουν προγράμματα αστικής κινητικότητας αν θέλουν να χρηματοδοτηθούν από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία. Ε, επίσης σε ένα δεύτερο σημείο και εδώ που δεν μας έχετε ακολουθήσει και κατ' εμέ ήταν ο για το, την πρώτη έκθεσή μου του σιδηροδρομικού πακέτου που είχαμε ζητήσει άπαξ και διαπιστώσαμε ότι το 60% των χρηματοδοτήσεων για τη συγχρηματοδότηση πηγαίνουν προς τις οδικές μεταφορές θα έπρεπε να επιστρέψουν στις σιδηροδρομικές μεταφορές και βεβαίως υπάρχει επικουρικότητα άρα αν θέλουμε να αλλάξουμε τις κλιματολογικές αλλαγές θα πρέπει να γίνει ε, κάτι διαφορετικό γι' αυτό και θα υποβάλω μία τροπολογία την οποία σας παρακαλώ να αποδεχτείτε γιατί είναι ο μοναδικός μοχλός το μοναδικό εργαλείο το οποίο έχουμε και τώρα εδώ δεν θέλω να πετάξω στον αέρα μη απαρίθμητα ε, μπαλόνια με αέρα κοπανιστό αλλά ε, νομίζω ότι θα πρέπει να ε, εκινήσουμε ορισμένα μπαλόνια διότι η Ευρώπη ποιείς ε, της πόλης ε, θα πρέπει ε, να βρίσκεται σε δεύτερη θέση. Οι πόλεις θα πρέπει να αποφασίσουν την ταχύτητα διακινήσεως μέσα στην πόλη και σε ποιους δρόμους θα μπορεί να πηγαίνει κανείς με 30 χιλιόμετρα. Δηλαδή, όπου υπάρχει μία διασταύρωση θα πρέπει να υπάρχει μία πινακίδα. Όπου υπάρχουν σχολεία και διαβάσεις θα πρέπει να υπάρχει υπάρχουν πινακίδες ε, για να μπορέσουμε να μειώσουμε και τα ατυχήματα και να βοηθήσουμε τις πόλεις. Αλλά οι πόλεις μπορούν να αποφασίσουν μόνες τους ποιοι είναι οι δρόμοι όπου μπορεί κανείς να κινηθεί με μεγαλύτερη ταχύτητα και πού όχι. Παρακαλώ λοιπόν να σκεφτείτε αν μπορούμε να έχουμε στο σημείο αυτό πλειοψηφία. Επίσης είπατε ευτυχώς ότι χρειάζεται ένας χάρτης για τους πεζούς ε, και είδαμε ότι ε, στην ε, Γερμανική μέρα των πόλεων μιλήσαμε και ε, για τις οδικές μεταφορές με ποδήλατο. Ε, λοιπόν, πολλές φορές βλέπουμε ότι οι ποδηλάτες δεν συμμορφώνονται με τις ενδείξεις των πόλεων και τις κρίνουν, αλλά κάποιος μου είπε ε, ότι υπήρχε τη δεκαετία του 80 ένας χάρτης για την κυκλοφορία των πεζών, την οποία θα μπορούσαμε να να αναβιώσουμε. Ε, και πέραν των πεζών πρέπει να μπορέσουμε να προστατεύσουμε και τους ποδηλάτες. Γενικώ όμως είμαστε ικανοποιημένοι με την έκθεση αυτή. Η εργασία ήταν καλή. Ευχαριστώ τον εισηγητή και παρακαλώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην ξανασυμπεριφερθεί όπως τώρα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπλόκλαντ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να, ε, ευχαριστώ, να ευχαριστήσω τον κύριο Σαβαρή για την εξαιρετική συνεργασία του και για το θαυμάσιο συντονισμό με τον οποίο συντάξαμε το κείμενο αυτό. Οπότε δεν χρειάζονται πάρα πολλά σχόλια παρόλο που υπάρχουν ορισμένες παρατηρήσεις ακόμη οι οποίες πρέπει να γίνουν διότι στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο δράσης για το περιβάλλον μας είχαν ε, υποσχεθεί 7 στρατηγικές. Τώρα υπάρχουν 6 ε, και εμείς περιμένουμε ακόμη μία στρατηγική για την περιβαλλοντολογική αστική πολιτική. Ε, είναι κάτι παρεμφερές με αυτά που συζητούμε εδώ. Ο κύριος Σαβαρή μίλησε για την κλιματολογική πολιτική που είναι του περιβάλλοντος. Υπάρχει επιπλέον και το πρόβλημα ε, των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακος αλλά υπάρχουν και οι βλαβερές εκπομπές ε, υπάρχει το θέμα της δημοσίας υγείας όλα αυτά λοιπόν μπορούν να συνδυαστούν και να καταρτιστεί μια καλή πολιτική των αστικών συγκοινωνιών που είναι κάτι που επιβάλλεται και παραμένει το θέμα της επικουρικότητος. Δηλαδή στην παράγραφο 14 ιδιαιτέρως ε, εκεί υπάρχει ουσιαστικά η κριτική μου διότι μήπως θα έπρεπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας κάνει μία έκθεση για τα διόδια στις πόλεις. Εγώ ανησυχώ, γιατί δεν ξέρω αν στα πλαίσια της επικουρικότητας μπορούμε να ζητήσουμε ένα μια τέτοια έκθεση. Αν την άλλη πλευρά είμαι πολύ ικανοποιημένο με τα ευέλικτα μέτρα μεταφοράς όπως το περπάτημα και το ποδήλατο. Θα μπορούσαμε ίσως να προσθέσουμε κάπου ότι αυτοί η τρόποι μεταφοράς είναι πολύ σημαντικοί. Θα έπρεπε δηλαδή να μπορεί κανείς να μεταφέρει ε, μέσα στο μετρό, στο λεωφορείο ή στο τραμ το ποδήλατό του. Ε, είναι μικρά θέματα, αλλά ε, πρόκειται για σημαντικά θέματα που ήδη έχουν αναφερθεί. Για τις πόλεις όπου υπάρχουν ήδη εμπειρίες μεταφοράς του ποδηλάτου μέσα στα μέσα μεταφοράς, θα είδαμε τις εντυπώσεις να είναι θετικές. Επίσης εδώ μιλάμε για πόλεις ε, πάνω των 250.000 κατοίκων και αλλού για 100.000 κατοίκους. Εγώ θα έλεγα λοιπόν στην παράγραφο 10 να μειώσουμε τους αριθμούς ε, των κατοίκων από 250.000 σε 100, πράγμα το οποίο είχαμε συζητήσει. Τελευταία παρατήρηση για την παράγραφο 12 όπου λέγεται ότι δεν θέλουμε ένα ε, νέο γραφείο. Μπορεί αυτό να λεχθεί ε, με περισσότερη στεναρότητα. Δεν θέλουμε καμία, καμία καινούργια υπηρεσία και καλό θα ήταν να το αναφέρετε με ε, περισσότερο στόμφο. Αυτά είχα να πω. Υπάρχουν ε, ορισμένες ε, μικρές προσθήκες, αλλά είναι μεγάλη χαρά μας να μπορούμε να παρουσιάσουμε κάτι τέτοιο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να το συζητήσουμε προτού αλλάξει η φρουρά και προτού αλλάξει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους αυτούς οι οποίοι συνεργάστηκαν για την έκθεση αυτή. Θα ήθελα όμως καταρχήν να πω ότι εγώ ε, είμαι από τα άτομα που δεν ικανοποιημένα με τις εσωτερικές μεταφορές μέσα στην πόλη και τις συγκοινωνίες. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπερεύει τις αρμοδιότητές της και ήταν ενάντια στην επικουρικότητα. Στα κράτη-μέλη όμως η κατάσταση διαφέρει από το ένα στο άλλο. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τα κράτη-μέλη μεταξύ τους. Εμείς δηλαδή έχουμε σε πόλεις που είχαν ισοπεδωθεί στον πόλεμο και τώρα οι δρόμοι είναι ίσως πιο φαργοί για τον αριθμό των αυτοκινήτων τα οποία κυκλοφορούν ενώ σήμερα το πρωί στις Βρυξέλλες χρειάστηκα για ένα σημείο 2 χιλιόμετρων μία ώρα ε, και αυτό βλέπετε περιγράφει πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση ε, της κυκλοφορίας της πόλης. Τώρα, ε, νομίζω ότι δεν υπάρχουν νέες αχθές αρχές. Ε, η κατάσταση των αστικών συγκοινωνιών μου θυμίζει την Ατζέντα 21, ε, την οποία είχαμε συζητήσει πριν από πολλά χρόνια δηλαδή πώς τα αστικά προβλήματα συγκοινωνίας μπορούν να επιληθούν και πώς μπορεί να υπάρχει ε, ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις βελτιώσεις. Δεν έχω τίποτα εναντίον του προγράμματος δράσης, αλλά είναι ε, πολυμορφικό και δεν ξέρω πώς θα μπορέσουμε έτσι ε, να προχωρήσουμε. Πολλά όμως έχουν ήδη ε, ρυθμιστεί. Υπάρχουν τεχνικές προδιαγραφές για τα λεωφορεία, για τα οχήματα. Έχουμε διάφορε θέματα που έχουν επιληθεί όπως είναι μέσω της οδηγίας για το θόρυβο, μέσω της οδηγίας για τα επίπεδα των εκπομπών και το ερώτημα είναι πάντοτε για την επικουρικότητα. Δηλαδή, εάν θέλουμε να εφαρμόσουμε ένα τέτοιο πρόγραμμα, είναι κάτι που πρέπει να, ε, να γίνει πολύ προσεκτικά. Οι στόχοι καταγράφονται επίσης. Αν δηλαδή ε, μπορούν τα θέματα αυτά να επιληθούν μέσω ενός ε, προγράμματος που θα περιλαμβάνει τις προτάσεις μας. Νομίζω ότι στην τελευταία ανάλυση πρέπει να αναλυφθεί από τις πόλεις που δεν έχουν χρήματα. Και αυτό είναι το πρόβλημα, διότι υπάρχει αστιφιλία και η αστιφιλία είναι κάτι που προωθείται για να μην καταστρέφουμε ε, και τα λιβάδια και από την άλλη πλευρά για να μην υπάρχει η μεταφορά από ε, ε, τα προάστια στην πόλη αλλά τότε οι πολίτες πολλές φορές δεν γνωρίζουν ότι καλύτερα θα ήταν να πηγαίνουν τις μικρές αποστάσεις με τα πόδια και να αφήσουν το αυτοκίνητο αυτοκίνητό του στο γκαράζ. Ε, θέλουμε, ε, θέλουμε επίσης να μην καταστρέψουμε το μικροεμπόριο στις πόλεις. Ε, έχουμε ένα πληθυσμό ο οποίος γερνάει όλο και περισσότερο και δεν μπορεί να πάει στα μεγάλα πολυκαταστήματα εκτός των πόλεων που είναι στην εξοχή για να κάνει τα ψώνια του. Δεν θέλουμε να καταστρέψουμε και το μικροεμπόριο, δεν θέλουμε να καταστρέψουμε το τοπίο εκτός πόλος, όλα αυτά λοιπόν ζητούν πολύ προσοχή. Επίσης όσον αφορά τις κατασκευές με το, τη, πολεοδομία, με τις δημογραφικές αλλαγές, όλα αυτά τα στοιχεία πρέπει να ληφθούν υπόψη διότι ε, η προσπάθεια είναι να επαναφέρουμε τον γυράσκοντα πληθυσμό στο κέντρο της πόλεως, να λύσουμε το πρόβλημα των μικρών μεταφορών ώστε οι άνθρωποι όπου μπορούν να κάνουν κάνουν τα ψώνια τους, όπου μπορούν να χρησιμοποιήσουν ε, δίκτυα μικρών αποστάσεων, ε, να μπορέσουν ε, να κινηθούν και εμείς να κάνουμε οικονομία πολλών συγκοινωνιών. Όλα αυτά όμως γίνονται χωρίς να σκεφτούμε το πολεοδομικό σχέδιο γενικώ. και το ερώτημα είναι πώς θα πρέπει να προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα διατυπώσει ένα πρόγραμμα δράσης. Επίσης Υπάρχει και το θέμα των ατομικών μεταφορών που και εγώ προωθώ. Είναι θέμα όμως οικονομικό. Το να ε, χρησιμοποιήσει κανείς ε, παραδείγματος χάρη το δικό του αυτοκίνητο εντός της πόλης είναι πολύ δαπανηρό διότι εγώ εάν θέλω να πάω δύο χιλιόμετρα έξω από την πόλη και πει ε, με το λεωφορείο η μία διαδρομή θα μου κοστίσει 2,5 ευρώ και μπορώ να το πληρώσω. Αλλά στην περιοχή μου που είναι μία παλιά βιομηχανοποιημένη περιοχή όπου υπάρχει μεγάλη ανεργία υπάρχουν πολλοί που δεν μπορούν να πληρώσουν κάτι τέτοια. Άρα τους είναι ε, φτηνότερο να πάνε με τα αυτοκίνητό τους αντί να πάρουν τα μέσα συγκοινωνίας. Επίσης ε, ε, υπάρχει θέμα ε, της, της μεταφοράς με ειδικού ποδηλατοδρόμους, με ειδικές διαδρομές για πεζούς για να μπορέσει να αυξηθεί το αίσθημα ασφαλείας των πολιτών, πράγμα το οποίο δεν πρόκειται να γίνει εάν κανείς φοβάται ότι θα του επιτεθούν τη νύχτα σε σκοτεινά σημεία της πόλης, οπότε ε, ε, ο προσωπικός τρόπος μεταφοράς δεν πολύ χρησιμοποιείται. Και τώρα θέλω ε, λίγο να αναφερθώ περισσότερο για, ουσιαστικά για την έκθεση σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για την προώθηση των δικτύων. Η πρόταση αυτή μου φαίνεται κάπως τολμηρή. Ε, είναι επίσης θέμα οικονομικό και εσωτερικής οργανώσεως των ε, επιχειρήσεων μεταφορών. Επίσης ε, προτείνεται να υπάρξει μία υπηρεσία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θεωρώ ότι είναι κάτι το περιττό διότι ήδη έχουμε ανταλλαγές σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ζητούμε να υπάρξουν ανταλλαγές ιδεών ε, και βελτίστων πρακτικών οπότε άπαξ και ζητάμε λύσεις ε, για τις μικρές αποστάσεις θα έπρεπε να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε κάτι τέτοιο δεν χρειάζονται νέες οργανώσεις, έχουμε επαρκής υπηρεσίας ε, και ξέρουμε ότι κάθε πόλη έχει το, το, το, τις δικές της οργανώσεις και αυτές πολλαπλασιάζονται. Επίσης όσον αφορά τη συγχρηματοδότηση των επενδύσεων για τους κοινοοικονομικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί από τον Ευρωπαϊκό Κορβανά, αυτό ε, ε, ούτως ή άλλως είναι εις βάρος αυτών οι οποίοι ήδη έχουν επενδύσει πολύ για να μπορέσουν να επιτύχουν πολιτικούς στόχους ενδεχομένως. Άρα δεν βλέπω γιατί το ποσοστό μας του ευρωπαϊκού ε, προϋπολογισμού πρέπει να διατεθεί τώρα στις πόλεις και εδώ είμαι πολύ αυστηρή. Πιστεύω ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να εξεύρουν μόνα τους αυτούς τους πόρους και μπορούν να υπάρχουν μεγάλες οικονομίες αφού προηγηθεί η ανταλλαγή των εμπειριών για να γνωρίζει ο καθένας πώς και μπορεί καλύτερα να επενδύσει. Αυτό που δεν βλέπω στην έκθεση και έτσι τελειώνω είναι το θέμα της εσωτερικής της μεταφοράς εντός των πόλεων των ε, ε, εμπορευματικών μεταφορών, ιδίως στις ώρες εχμής. Ε, διότι αυτή είναι η ώρα στην οποία παραδίδονται ε, και γίνεται η διανομή στο, κέντρο των πόλεων είναι κάτι το οποίο χρήση βελτιώσεως και αυτό που θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό θα ήταν ε, η έρευνα για την καλύτερη διανομή των εμπορευμάτων στο κέντρο της πόλεως. Νομίζω Νομίζω αυτό θα ήταν ε, μια πολύ αξιέπαινη προσπάθεια για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε σωστά τους ευρωπαϊκούς πόρους και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να συμφωνήσω με κάποιους ε, συναδέλφους που εξέφρασαν την απογοήτευσή τους όσον αφορά τη στάση της Κομισιόν. Όντως, η υπόσχεση που μας δόθηκε πολλές φορές κατά τη διάρκεια των δύο ετών για την ε, σχέδια δράσης είναι κάτι το οποίο δεν έγινε πραγματικότητα. Όντως, άκουσα ότι η Κομισιό για την αστική κινητικότητα σκέπτεται τα επόμενα χρόνια να κάνει κάτι. Το ελάχιστο μπορεί να κάνει είναι αυτό, θα έλεγα. Εμείς όμως θα θέλαμε ένα σχέδιο δράσης συνεκτικό και λογικό, στο οποίο θα απαριθμίζεται με συγκεκριμένο τρόπο τι προβλέπει να κάνει η Κομισιόν το 2009-2010 και τα επόμενα χρόνια. Γι' αυτό είναι κάτι το οποίο θα συνεισφέρει στην ορατότητα του τι κάνει η Ευρώπη, στην καλή κατανόηση πολιτικής και στο τι επιθυμούμε. Γιατί λοιπόν γίνεται κάτι, ποιος είναι ο στόχος. Όλα αυτά αρνείται να τα κάνει η Κομισιόν. Γι' αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή μας, τον συνάδελφο Σαββανή, που πήρε την πρωτοβουλία να μας παρουσιάσει ο ίδιος μία σχετική με τα θέματα αυτά έκθεση. Συμφωνούμε όλοι στο ότι Όντω υπάρχουν χίλιοι λόγοι που θα μπορούσαμε να μα να μιλήσουμε για την αστική κινητικότητα στι πόλει τη Ευρώπη. Δεδομένου τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε όλοι με τι μεταφορέ στην Ευρώπη είναι πολλά. Πιστεύω λοιπόν ότι το θέμα της επικουρικότητας θα πρέπει να το εκμεταλλευτούμε και να το συζητήσουμε σωστά με πνεύμα λογικής θα πρέπει να δούμε πώς μπορεί η Ευρώπη βοηθήσει τις πόλεις ώστε να βελτιωθεί η αστική κινητικότητα. Πιστεύω ότι μπορεί η Ευρώπη να τις βοηθήσει τις πόλεις αυτές και τότε θα πρέπει οι πόλεις να δώσουν συνέχεια στις ε, συστάσεις που θα γίνουν εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εξάλλου πάρα πολλά στοιχεία από αυτά περιλαμβάνονται στην έκθεση αυτή, δεδομένου ότι η Ευρώπη παίζει σημαντικό ρόλο στην έρευνα και στην ε, ανάπτυξη και χρησιμοποίηση νέων τεχνολογιών ώστε να έχουμε δημόσιες συγκοινωνίες πιο καθαρές και πιο αποτελεσματικές. Πιστεύω ότι η Ευρώπη μπορεί εύκολα να θεσπίσει και διάφορους κανόνες και προδιαγραφές για καθαρές μεταφορές, για καθαρές πόλεις και να παρουσιάσει διάφορους κανόνες και μέτρα για να βελτιωθούν τα πράγματα. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα μέσο, ένα παρατηρητήριο, κάτι το οποίο θα ανάλαβε τα θέματα. Δεν θέλουμε ένα νέο γραφειοκρατικό οργανισμό, αλλά μία, ε, ένα κέντρο, αν θέλετε, στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται όλες αυτές οι πρωτοβουλίες. Και επίσης να βρεθούν νέοι μηχανισμοί χρηματοδότησης ή να διορθωθούν κάποιες παρούσες ε, χρηματοδοτικές δράσεις για να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι το αποδοτικό. Πιστεύω ότι δεν χρειάζεται να λυθούν πάρα πολλές πρωτοβουλίες, αλλά οι σωστές που θα επιτρέψουν σε όλους να επομιστούν τις ευθύνες τους από το τοπικό, το κρατικό έως το κοινοτικό επίπεδο. Αυτά θα ήθελα να πω και τελειώντας και πάλι να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τον εισηγητή για την εργασία που επιτέλεσε. Γι' αυτό και τους συναδέλφους και πιστεύω ότι όλοι μπορούμε να στείλουμε ένα θετικό σινιάλο προς τα έξω. Ελπίζω ότι θα μπορέσει να πει κάτι η Κομισιόν και να αλλάξει γνώμη, να συμπληρώσει τις ε, πρωτοβουλίες μας και να κάνει κάτι το χρήσιμο. Ευχαριστώ κυρία Κικάου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ τον εισηγητή μας τον κύριο Σαβαρή για την άριστη δουλειά του. Τότε υπάρχει ομοφωνία εκ μέρους των σχεδόν εισηγητών είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τη συζήτηση. Όσον αφορά την αστική κινητικότητα, πρέπει να μιλήσουμε για τον προγραμματισμό για τις πόλεις, δηλαδή πώς θα κτίζονται στο μέλλον οι ευρωπαϊκές πόλεις και ποιος θα είναι ο ρόλος της υποδομής μεταφορών επίσης το πώς συνδέονται οι διάφοροι τρόποι μεταφοράς. Δηλαδή να μπορεί να φτάνει κανείς στο αεροδρόμο με μετρό ή με ένα γρήγορο τρένο χωρίς να είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιήσει τις οδικές μεταφορές. Γιατί υπάρχει ένας κώδικας που υπολογίστηκε για τη συμφόρηση 1% του ΑΕΠ της Ένωσης του ΑΕΠ. Αν έχουμε εναλλακτική χρήση διαφόρων μέτρων μεταφοράς, αυτό το κόστος μπορεί να μειωθεί. Παρακαλώ τον κύριο Σαβαρή στην έκθεσή του να βάλει και μερικά στοιχεία για την ασφάλεια. Γιατί όλοι όσοι παίρνουν μέρος, όσοι συμμετέχουν στο σύστημα αυτό των μεταφορών, θα πρέπει να ε, καλύπτονται από προστασία. Δηλαδή, ε, επίσης κάτι άλλο, πρέπει να προωθηθούν τα δημόσια μέσα μεταφοράς, είτε χρησιμοποιώντας έξυπνα συστήματα μεταφοράς, είτε ενσωματώνοντας τις διάφορες μορφές δημόσιων μέσων μεταφοράς και ειδικά τα έξυπνα συστήματα στις μεταφορές θα είναι χρήσιμη για καλύτερη χρήση αυτών των μέσων. Είναι χρήσιμο κάπως κάποιος να μπορεί να υπολογίζει στο ωράριο των μέσων μεταφοράς, το οποίο να τηρείται. Σχετικά πρόσφατα στο Κοινοβούλιο εγκρίθηκε μια οδηγία που αφορά τα καθαρά οχήματα. Δεν μιλάμε πολύ για αυτή την οδηγία. Στην πράξη η τοπική αυτοδιοίκηση έχει τη δυνατότητα όταν αγοράζει ένα λεωφορείο ας πούμε για τις συγκοινωνίες να μπορεί να υπολογίσει την κόστο χρήσης για όλη τη διάρκεια ζωής του λεωφορείου. Όχι μόνο που τους τύχησε να το αγοράσουν, τις εκπομπές και λοιπά όλα. Ελπίζω αυτή εδώ η έκθεση να αποτελέσει τη βάση για μια αναθεώρηση των διορθωτικών ταμείων του 2010 εννοώ. Οπότε θα υπάρχει η δυνατότητα να βάλουμε νέες προτεραιότητες, να κάνουμε συστάσεις προς τα κράτη-μέλη για να έχουμε καλύτερη απορρόφηση των διορθωτικών κονδυλίων. Πιστεύω ότι η αστική κινητικότητα μπορεί να είναι τέτοια προτεραιότητα. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Ένα λεπτό. Ναι, ε, οι πόρες έχουν ε, αλλάξει και έχουν επηρεαστεί ε, διαφορετικά από τον πόλεμο αλλά πολλές φορές άφησαν τον χώρο πάνω από τη γη για τα, αυτοκίνητα και χρησιμοποίησαν τον υπόγειο χώρο για το μετρό. Όταν λοιπόν λέμε ότι χρειαζόμαστε αυτοκίνητα για να μπορέσει να υπάρξει υπάρξει εμπόριο στο εσωτερικό των πόρων δεν είναι σωστό θα πρέπει να υπάρχει ούτως ή άλλως και ο ανταγωνισμός εκ των έξω. Δυστυχώς το μικρόφωνο του ομιλητή δεν λειτουργεί πλέον. Και στη Βενετία το κάναμε το ίδιο. Η κυρία Ότμαν της Κομισιόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. όπως απέδειξε η συζήτηση, η διαβούλευση μετά το πράσινο βιβλίο για την αστική κινητικότητα απέδειξε ότι υπήρχε αρκετά μεγάλη συμφωνία μεταξύ ενδιαφερομένων για το ότι μπορεί να διαδραματίσει ρόλο σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια της αρχής της επικουρικότητας. να σας πω σήμερα, σε σχέση με τη διαβούλευση, ότι υπάρχει η σχετική διάσκεψη που λαμβάνει τώρα σήμερα και από σήμερα δημοσιεύονται τα αποτελέσματα στο σχετικό site της Επιτροπής. Όπως είπε και ο εισηγητής, ο στόχος της προσυνοβιβλίου ήταν να προετοιμαστεί το έδαφος για να υπάρξει σχέδιο δράσης για την αστική κινητικότητα που ακόμη δεν έχει εγκριθεί. Παρ' όλα αυτά, ο Αντιπρόεδρος Ταγιάννη πολλές φορές επιβεβαίωσε από τότε ότι αναλαμβάνει αποφασιστικά δράση ώστε στο εγγύς μέλλον να υπάρξει ενσωματωμένο και ευρύτερο σχέδιο δράση. Το σχέδιο δράση αυτό βρίσκεται και στο πρόγραμμα εργασίας της Κομισιόν για το 2009. Ακόμη όμως και αν δεν υπάρχει σχέδιο δράσης, πρέπει να σας πω ότι η Επιτροπή συνεχίζει τις δράσεις της κάποιες από τις οποίες ήδη θα τεθούν σε κίνηση φέτος. Την προηγούμενη εβδομάδα, στην τοποθέτησή της για την έκθεση Φλόρενς που αφορά τις κλιματικές αλλαγές, η Κομισιόν υπενθύμησε τις δεσμεύσεις της να αναπτύξει δράσεις στον τομέα της αστικής κινητικότητας και αυτή τη στιγμή, όπως είπα, λαμβάνει χώρα μία διάσκεψη για την αστική κινητικότητα που οργάνωσε η Κομισιόν, στην οποία συμμετέχουν 350 άτομα εκ από όλη την Ευρώπη για να συζητήσει ε, κάποια θέματα και πρωτοβουλίες που αφοράν ε, τις ε, οικολογικές ε, ε, κρατικές προμήθειες, κάποιους δημόσιους χώρους, κάποια άλλα θέματα και επίσης τα μεταβιώσιμων ενεργειών για να μπορέσουμε να λάβουμε συγκεκριμένες μέτρα. Η πρωτοβουλία σας, εσείς, να δημιουργήσετε το δικό σας σχέδιο δράσης στα πλαίσια αυτή τη πρωτοβουλία, δεδομένου ότι δεν έχει κάνει τίποτα μέχρι τώρα η Κομισιό, είναι σημαντική διότι στέλνει ένα πολύ σημαντικό πολιτικό μήνυμα. Αποδεικνύει ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες που εκπροσωπεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναγνωρίζουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να διαδραματίσει ρόλο και αναμένουν δράσεις εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σχέδιο έκθεσης του κυρίου Σαββαρή επιβεβαιώνει ότι η στική κινητικότητα είναι μέρος όντως της κοινή πολιτικής μεταφορών. Ο ρόλος αυτός επιβεβαιώνεται εξάλλου και στο πράσινο βιβλίο για τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών, τα οποία ενέκρινε η Επιτροπή και θα επιβεβαιωθεί εξάλλου και στην ανακοίνωση που θα παρουσιάσουμε τον Ιούνιο για το μέλλον των μεταφορών μακροπρόθεσμα. Η έκθεση που προτείνεται εδώ συμπεριλαμβάνει έναν φιλόδοξο κατάλογο πολύ καλά στοχευμένων προτάσεων που αναμφίβολα έχουν μία προσθέμενη αξία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχει μεγάλη σύγκληση απόψεων με τις προπαρασκευαστικές εργασίες που κάναμε εμείς σε επίπεδο Επιτροπής για το σχέδιο δράσης και το σχέδιο έκθεσης αυτό σίγουρα αποτελεί μια πάρα πολύ χρήσιμη συνεισφορά στις εσωτερικές συζητήσεις που κάνουμε για την ολοκλήρωση του σχεδίου δράσης της Κομισιόν. Μπορούμε να εμπνευστούμε από πολλές από τις προτάσεις που περιλαμβάνονται και θα το κάνουμε αυτό. Ο πραγματικός περιορισμός που έχουμε εμείς είναι πραγματικά η έλλειψη κονδυλίων και οικονομικών και σε ανθρώπινο δυναμικό. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Γκούτμαν, διότι μας ε, έδωσε κάποιες διαβεβαιώσεις όσον αφορά τις προθέσεις επιτρούς και διότι μας ενθάρρει να συνεχίσουμε, δεδομένου ότι τώρα έχουμε μπει σε ένα κλίμα αμοιβαίου επηρεασμού ημέν των δε πράγμα, το οποίο πιστεύουμε ότι θα οδηγήσει σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράση εκ μέρους Κομισιόν. Σίγουρα για την επόμενη θητεία. Δεν ήθελα να απαντήσω στους συναδέλφους να πω ότι συμφωνώ λαμβάνω υπόψη διαφορετικές παρατηρήσεις που έγινε, θέλω να στον κύριο Κράμερ ότι εάν δεν ενσωμάτωσα το 40% της χρηματοδότησης για τις συνδρομικές μεταφορές είναι διότι δεν θέλησα να ε, υιοθετήσω μία προσέγγιση πάρα πολύ ε, ε, η οποία θα δημιουργεί υποχρεώσεις θα μπορούσε να μας να οδηγήσουν κάποιον να πούμε ότι την παίρνουμε στα χωράφια άλλους. Ξέρουμε ότι κάποιες, ε, για τις δρομικές μεταφορές, κάποιες ε, πόλεις ε, προσφέρονται, κάποιες άλλες όχι και θα πρέπει ίσως σε αυτή την περίπτωση να προωθηθεί περισσότερο το σχέδιο δημιουργίας περισσότερων προσδρόμων ή άλλων τόπων ειδικών. Εντάξει, δεν θα κάνουμε εμείς πολιτική στο επίπεδο των πόλεων, τους αφήνω του υπεύθυνου να το κάνουν. Και δεν θέλω βεβαίως μέσα στην ε, έκθεση να βάλουμε πάρα πολύ αντιφατικές προτάσεις για να μας, μη μας ε, κατηγορήσει κανείς ότι θέλουμε να υποστηρίξουμε τις ειδικές Το βαπορέτο λοιπόν δεν θέλησα να το συμπεριλάβω, παρόλο που είναι περιορισμένη. Εσείς κύριε Πρόεδρε. Κύριε Μπλόκλαντ, λαμβάνω υπόψη παρατηρήσεις που κάνατε για τα θέματα δημόσιας υγείας. Εγώ είμαι της γνώμης ότι θα πρέπει να ενεργήσουμε και στα πλαίσια των ενεργειών που γίνονται την προσέγγιση του περιβάλλοντος, αλλά όχι μόνο. Θέλουμε να βελτιώσουμε το αστικό περιβάλλον για να βελτιωθεί και η δημόσια υγεία, κυρίως οι διάφορες πνευμονικές παθήσεις. Τώρα, στο σημείο 14 είναι εδώ για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα διότι πιστεύω ότι είναι ένα μέσο το οποίο θέλουν να, θεσ... να διαθετήσουν ε, διάφορες πόλεις και πιστεύω ότι είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να βοηθήσει διάφορες πόλεις, τη οχώνει και κάποιες άλλες και επίσης τα οδικά ε, διόδια στα αστικά κέντρα είναι κάτι το οποίο είναι πολύ ειδικό για κάποιες πόλεις. Θα θέλαμε λοιπόν να ξέρουμε ποιες είναι οι επιπτώσεις στην, ε, όσον αφορά την ε, ανταγωνισμό που υπάρχει μεταξύ των διαφόρων άλλων μέσων μεταφοράς. Όπως είπαμε, θέλουμε να, δοθεί, να δοθούν κίνητρα ώστε να υπάρξει προγραμματισμός των αστικών διαφορετικών συγκοινωνιών της Ευρώπης. Είπαμε ότι θέλουμε ένα κατόφλι πόλεων 250.000 κατοίκων. Θέλουμε εμεί να δημιουργήσουμε κίνητρα στους υπεύθυνους όλα αυτά εξαρτώνται και από τη δομή του κάθε κράτους. Στη Γαλλία για τις αστικές συγκοινωνίες σε κάποια αστικά κέντρα είναι υπεύθυνη η τοπική αυτοδιοίκηση για τα διάφορα υπεραστικά, αν θέλετε, για τις διάφορες υπεραστικές συγκοινωνίες είναι υπεύθυνοι κάποιοι από την νομαρχία, αν θέλετε, όπως τα λέγαμε σε επίπεδο ελληνικό, κάποιοι από το δημοτικό διαμέρισμα, από το νομό, τέλος πάντων. Θα θέλαμε λοιπόν να υπάρχει σωστή οργάνωση εκ μέρους όλων για να βελτιωθεί η κατάσταση. Όσον αφορά το παρατηρητήριο, νομίζω ότι πρόκειται για μια δομή αρκετά ελαφρά που θα πρέπει κυρίως ε, να τροφοδοτήσει την ανταλλαγή βελτίστων πρακτικών. Αλλά πρέπει να τις έχει κανείς για να τις ανταλλάξει αυτές τις βέλτιστες πρακτικές. Όσον αφορά τον προπολογισμό, Λαμβάνω υπόψη αυτό που ελέγχθη για να δοθεί περισσότερη υποστήριξη στα θέματα μεταφορών φρέτ, δηλαδή των εμπορευμάτων εντό των πόλεων. Μπορούμε νομίζω εδώ να πούμε κάτι περισσότερο σχετικά αφορά τα κονδύλια που θα πρέπει να ε, δοθούν, αν θέλουμε να δημιουργήσουμε κίνητρα, βεβαίως θα πρέπει να διαθέσουμε και πόρους. Ο προϋπολογισμός 2013-2020 ξέρω ότι θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένες σε νέες ανάγκες της και ξέρω ότι υπάρχουν περιορισμοί. Έχουμε νέε επιταγέ, νέε ανάγκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά εάν θέλουμε να προωθήσουμε την προστασία του κλίματος, να μειώσουμε τα φαινόμενα εκπομπόκας και δηλαδή δημιουργία ε, των αερίων θερμοκηπίου θα ε, πρέπει κάτι να κάνουμε. Δεν ξέρω πώς θα το ονομάσουμε, τον Τζέκις Χάν, κάπως για τις αστικές συγκοινωνίες, για να μπορέσουμε να προωθήσουμε τους καλύτερους δυνατούς τρόπους. Τελειώνοντας, θα ήθελα να πω ότι χαιρετίζουμε το ότι υπάρχουν τα αποτελέσματα του πράσινου βιβλίου. Θα τα εξετάσουμε με μεγάλο ενδιαφέρον και πρέπει να πω ότι στα πλαίσια της μας πρωτοβουλίας όσοι ενδιαφέρονται από το θέμα αυτό μας έδωσαν ε, τα πορίσματα στα οποία κατέληξαν είχαν χτυπήσει ή κατάλαβαν λάθος πόρτα, έφυγαν την Κομισιό, ήρθαν σε εμά, συνεισέφεραν ε, πολύ στις δικές μας παρατηρήσεις και κρίσεις. Σου ευχαριστώ και θα ήθελα όντως εγώ να πω ότι η πολιτική μας προσέγγιση για να ψηφιστεί η έκθεση αυτή τον Απρίλιο θα θέλαμε να οδηγήσει στην ύπαρξη ενός σχεδίου δράσης για την αστική κινητικότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι η κατάλληλη στιγμή, είναι επίκαιρο το θέμα και την ε, στιγμή κατά την οποία εμείς ε, θα χρειαστεί να ακυρώσουμε τον ορισμό των νέων ε, επιτρόπων, καλό θα είναι να έχουμε κάνει αυτή τη δουλειά. Προτείνω προθεσμία κατάθεση τροπολογιών τη 18η, διότι όπω είπαμε θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το χρονοδιάγραμμα. Ε, δεν έχουμε πολύ χρόνο, σα δίνω μια εβδομάδα καιρό. Και εάν εγώ ε, δω ότι πρέπει να καταθέσουν κάποιε τροπολογίε, θα τι ε, στείλω στου σκιώδει ε, εισηγητέ, ώστε να μπορέσουμε να επιταχύνουμε την όλη διαδικασία. Σα ευχαριστώ πολύ για την συνεργασία και τη συνεισφορά σα στην συζήτηση τη σημερινή. Πρόεδρος, έχουμε μία εβδομάδα για τι τροπολογίες μέχρι 18 Φεβρουαρίου για να τη ε, ψηφίσουμε το κείμενο τον Μάρτιο και να πάμε στα λομέλια τον Απρίλιο. Πέρας συνεδρίασης. ΟΚ. Okay, okay.